Diamo inizio. Shall we start? Σας ευχαριστώ. Ε, παρακαλώ να καθίσετε να ξεκινήσουμε. Benvenuti, benvenuti cari colleghi. Καλώς ορίσατε Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε και σε όσους επανέρχονται στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξη Πέθρου και καλώς ορίσατε και σε όσους ε, νέους συναδέλφους ήρθαν σε αυτή τη σημαντική Επιτροπή. Όπως γνωρίζετε σήμερα, η συνεδρίασή μας θα αναμεταδίδεται στο διαδίκτυο και θα υπάρχουν όλες οι γλώσσες διαθέσιμες και 23 Η σημερινή συνεδρία, όπως γνωρίζετε, είναι αφιερωμένη στη σύσταση της Νέας Επιτροπής. Άρα λοιπόν πρέπει να εκλέξουμε τον νέο πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας. Μετά θα γίνουν εκλογές για τους τέσσερις αντιπροέδρους της ίδιας Επιτροπής. Νομίζω πως τώρα είναι σκόπιμο να θυμίσω σε όλους σας ότι Εάν υπάρξουν περισσότερες από μία υποψηφιότητες θα πρέπει να ψηφίσουμε με την κάρτα ψηφοφορίας. Γι' αυτό σας παρακαλώ όλους να έχετε έτοιμη την κάρτα ψηφοφορίας σας, εάν τυχόν χρειαστεί να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Συνάδελφοι, λοιπόν, πρέπει τώρα να προχωρήσουμε στην εκλογή του Προέδρου. Να είναι επειδή εγώ θέλω να μείνω πρόεδρος, γι' αυτό έκανα λάθος και είπα για αντιπρόεδρος κατευθείαν. Να σας θυμίσω ότι το γλωσσικό προφίλ έχει αφαιρεθεί από την ημερήσια διάταξη, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στην εκλογή του νέου Προέδρου. Συνάδελφοι, Να ξεκινήσω με τη διαδικασία και να θυμίσω σε όλους ότι έχουμε λάβει την υποψηφιότητα του συναδέλφου Σικέρσκη. Καταρχήν να ρωτήσω τον συνάδελφο Σικέρσκη εάν τι δέχεται αυτή την υποψηφιότητα. Yes, ε, Μάλιστα. Και τώρα πρέπει να ρωτήσω εάν υπάρχουν άλλοι υποψήφοι. Αν κάποιος άλλος συνάδελφος θέλει να υποβάλει υποψηφιότητα κάποιου άλλου ε, συναδέλφου για προεδρία της Επιτροπής. Μάλιστα. Εφόσον δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος, μπορούμε να εκλέξουμε το συνάδελφο Σικέρσκι, πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξη Πέθρου, διαβοής. Συγχαρητήρια. Και τώρα, αγαπητέ Σεκέρσκι, έλα ε, στο Προεδρείο να πάρει τη θέση μου, όχι πλέον ως Αντιπρόεδρος, αλλά ως Πρόεδρος της Επιτροπής. Και καλή επιτυχία από πλευράς μου και καλή δουλειά. Dziękuję panu przewodniczącemu De Castro za przeprowadzenie Ευχαριστώ κύριε Σας ευχαριστώ όλους που με εκλέξατε πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας. Ευχαριστώ και τον πρόεδρο, τον Πελθόντα, Κάστρο και όλους εσάς. Επειδή δεν έχουμε όμως πολύ χρόνο, να περάσουμε στο επόμενο σημείο της διάταξης, που είναι η εκλογή των αντιπροέδρων της Επιτροπής Άγκρη. Przechodzimy. Jeszcze raz serdecznie Państwa witam. Προχωρούμε λοιπόν. Σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στην ε, συνεδρίαση. Και περνάμε στο επόμενο σημείο της μέρης διάταξης. Αν έχετε διαβάσει τον εσωτερικό κανονισμό, θα γνωρίζετε ότι μετά την εκλογή του Προέδρου πρέπει να εκλέξουμε τους αντιπροέδρους Επιτροπής. Γεωργίας και θα ψηφίσουμε χωριστά τον ένα μετά τον άλλο. Εκλογή πρώτου αντιπροέδρου. Υπάρχουν υποψηφιότητες. Προτείνω ως πρώτη, πρώτη την Τζούλια Μόη. Ευχαριστώ, κύριος Άγγνιου ήταν. Σας ευχαριστώ κύριε Άγνου Ο κύριος Δεκάστρο θέλει το λόγο, παρακαλώ. Πρόεδρε, εγώ εξ ονόματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατικών προτείνω τον συνάδελφο Ερίκ Αντρέ ως πρώτο αντιπρόεδρο αυτής της Επιτροπής. Υπάρχουν άλλοι υποψήφοι. Όχι. Οπότε παρακαλώ. Στρέφομαι στους δύο υποψηφίου. Και τους ερωτώ, συμφωνείτε με την υποψηφιότητα κυρία Μόη καταρχάς. Συμφωνείτε με την υποψηφιότητα. Συμφωνείτε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντρίε. Oui, Ναι, βεβαίω, συμφωνώ. Κυρίε και κύριοι, θέλω τώρα να προτείνω να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Έχετε όλοι τις κάρτες σας. θα ψηφίσουμε ως εξή. Όλοι, είτε τακτικά μέλη, είτε αν τους αντικαθιστά ένας αναπληρωτής μπορούν να ψηφίσουν, έχουν δικαίωμα μίας ψήφου ο καθένας. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στην ψηφοφορία. you have to read the list of substitutes. Mm -hmm. You have to, to read it. Mm-hmm. Chcę, chcę Państwa poinformować, że... Θα ήθελα να σας πω ότι ο κύριος Κώστηκα αντικαθίστα τον κύριο Λίντς, ο κύριος Καρινόσκι από την κυρία Αγιούσο, ο κύριος Μέλα και Ακανιέτα. Επίσης, Γκαρθία Πέρες αντικαθιστά την κυρία Γκίλαρ. Να δώσω το λόγο στον συνάδελφο. Εμεί, η αποτελική μα πολιτική ομάδα, λαμβάνει, χώρα, ε, λαμβάνει μάλλον μέρο στην ψηφοφορία ο κ. Μπουβέ. Και εγώ αντικαθώ τον κύριο Όντε, λέει ο κύριος Ολιρέν. Ωραία, σας ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, διευθετήσαμε το θέμα των αναπληρωματικών και μπορούμε να περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία. Θα σας εξηγήσω πώς θα διεξαχθεί η ψηφοφορία. Αν θέλετε να ψηφίσετε τον κύριο Άντριε, πατάτε το πράσινο κουμπί. Εάν θέλετε να ψηφίσετε τον άλλο υποψήφιο, την άλλη υποψήφιο, πατάτε το κόκκινο και αν θέλετε να απόσχετε πατάτε το λευκό. Αλφαβητικά δηλαδή αναφέρω τους υποψηφίους. Άντριε πράσινο, μόι κόκκινο. Όποιος θέλει να απέχει πατάει το λευκό κουμπί. Αν είναι σαφές για όλους, μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. έναρξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τον πρώτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής μας. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα με το μηχάνημα, δυστυχώς κύριε Πρόεδρε. Εντάξει. Υπάρχει κάποιος άλλος που έχει πρόβλημα με το μηχάνημα. Όχι. Ωραία. Αν είναι να μην ενημερώσετε παρακαλώ ένδειξη ψηφοφορία, λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Με ενημερώνουν ότι από τους σοσιαλιστές ψηφίζει ένας παραπάνω. Κάποιος λοιπόν πρέπει να βγάλει την κάρτα. Πρέπει να το διορθώσουμε αυτό. Οπότε πρέπει να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Επειδή πριν ήταν ένας σοσιαλιστής περάριθμος. Έναρξη της ψηφοφορίας. Γέννη. Ψηφίζεται. Υπάρχει κάποιος ε, που να αντιμετωπίσει πρόβλημα με το μηχάνημα. Όχι. Λοιπόν, πέραση ψηφοφορία. Πέραση, επαναλαμβάνω, τη ψηφοφορία. Ο κύριος 27 ψήφους, η κυρία Μόη 8. Είχαμε και 5 αποχές. Επομένως, Πρώτος αντιπρόεδρος εκλέγεται ο κύριο Αντριέ. Συγχαρητήρια. Παρακαλώ τον πρώτο αντιπρόεδρο να έλθει εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Μόη, τη δεύτερη υποψήφια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι. Και τώρα προχωρούμε στην εκλογή του δεύτερου αντιπρόεδρου. Υποψηφιότητες, παρακαλώ, κύριε Νίκολσον. Ναι, κύριε Πρόεδρε, προτείνω τον κύριο Γιάννου Βαντιτσκόφσκι που ήταν τα προηγούμενα δυόμιση χρόνια αντιπρόεδρος Επιτροπής. Γιάννους Pan poseł Janusz Wojciechowski. Δέχεστε. Δέχομαι. Ο κ. Ντες. Ευχαριστώ. Ο κ. Γιάννα Διεργία Σάιερ. Ωραία, το σημειώνουμε αυτό. Καταγράφεται. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλοι υποψήφοι. Θα πρότεινα λοιπόν να κλέξουμε διαβοή στον κύριο Βοτσυχόσκη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Βοητσεχόσκι, να έλθει παρακαλώ στο Προεδρείο. Περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία, αφού συγχαρώ τον κύριο Βοητσεχόφσκι. Περνάμε στην εκλογή του τρίτου αντιπροέδρου της Επιτροπής Γεωργίας. Υποψηφιότητες παρακαλώ, η θέση του τρίτου αντιπροέδρου. Υποψήφοι παρακαλώ υπάρχουν για τη θέση του τρίτου αντιπροέδρου. Ο κύριος Δεκάστρο έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να υποδείξω ω τρίτο αντιπρόεδρο τη συνάδελφο Αγγιλάρ Γκαρσία Κλάρα, εξ ονόματος ε, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Στεφόμαι το στην υποψήφια. Δέχεται Κύριε έχετε πάλι το λόγο. Κοιτάξτε, δυστυχώς η συνάδελφος Αγγιλάρ δεν είναι παρούσα, αλλά γραπτός ε, εξέφρασε την αποδοχή της υποψηφιότητας της για την τρίτη την Προεδρία. Ωραία. Είναι παραδεκτή η γραπτή αποδοχή. Υπάρχουν άλλοι υποψήφοι για τη θέση αυτή. Έχουμε άλλη μία υποψηφιότητα. Θέλετε το λόγο κύριε Άγνιο. Ο κύριος Άγνιο. Εγώ θα προτείνω τον κύριο Ζόλε της ομάδας EFD για την θέση του τέταρτου αντιπρόεδρου της ε, κοινοβουλευτικής, του τρίτου συγγνώμη, του τρίτου αντιπρόεδρου της κοινοβουλευτικής επιτροπής. Παρεμβάσεις αλλά χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς. Mm-hmm. Euh, euh, ευχαριστώ κύριε Ζόλο. Είστε τακτικό μέλος της Επιτροπής. Μπορείτε λοιπόν να είστε υποψήφιος για το αξίωμα αυτό. Είστε διατεθειμένος να κατέρχεται υποψήφιος. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Έχει καλός, ο πρόεδρος κ. Σικιέσκη. Ας προχωρήσουμε λοιπόν τότε σε ηλεκτρονική ψηφοφορία με, αλφαβητικό, με αλφαβητική σειρά. Επομένως πρώτα η κυρία Αγγιλέρα Γκαρσία για το πράσινο κουμπί λοιπόν, με το πράσινο κουμπί και ο κύριος Ζούλο κόκκινο κουμπί. Είναι σαφές και κατανοητό για όλους και όλους. Αν συμφωνείτε λοιπόν τότε ας προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Παναλαμβάνω το ονόμα των δύο υποψηφίων. Αγγιλέρα Γκαρσία, ε, τότε πατάτε το πράσινο κουμπί. Εάν επιθυμείτε να ψηφίσετε υπέρ του κυρίου Ζούλο, το κόκκινο. Αρχίζει η ψηφοφορία. Oui, fermé. Νομίζω τώρα ότι μπορούμε να κλείσουμε την ψηφοφορία. Δεν σημειώθηκαν τεχνικά προβλήματα. Επομένω εδώ λίγη η ψηφοφορία. Η κυρία Αγγιλέρα λαμβάνει 24 ψήφους, ο κύριος Ζούλο 11. Άρα εκλέγεται η κυρία Κιλέρα Γκαρσία στην θέση της τρίτης αντιπροέδρου, εν απουσία της, αλλά βεβαίως ευχαρίστως να προσέλθει στο Προεδρείο την επόμενη φορά. Τώρα θα προχωρήσουμε στην ε, εκλογή του τετάρτου αντιπροέδρου. Υπάρχουν υποψηφιότητε για την θέση του τετάρτου αντιπροέδρου. Κύριε Δεκάστρο, εσείς πάλι. Μάλιστα, Πρόεδρε, εγώ θέλω να ανακοινώσω την υποψηφιότητα της κυρίας ε, Ντάντσιλα Μπαζίλικα, εξ ονόματος Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ο Πρόεδρος, κ. Σικέρσκη. Ο Πρόεδρος, κ. Σικέρσκη. Η κυρία Βασίλικα ενδιαφέρεται να κατέρθει υποψήφια. Μάλιστα, συμφωνώ. Υπάρχουν άλλοι ή άλλες υποψήφοι. Άγνιο. Θα ήθελα, εάν είναι δυνατό, να προτείνω την ίδια υποψηφιότητα όπως προηγουμένως. Προτείνω λοιπόν και πάλι την Τζούλια Μόη για, το τέταρτη, τη θέση του τέταρτου του Προέδρου της ε, Επιτροπής. Η γραμματεία μου εξηγεί ότι είναι δυνατό. Η κυρία Μόη θέλει όντως να ε, είναι υποψήφια. Μάλιστα. Επομένως έχουμε πάλι δύο υποψηφίους. Μάλιστα δύο υποψήφιες. Πολύ ωραία. Ας ψηφίσουμε λοιπόν, ξεκινώντας πάλι αλφαβητικά, Πρώτη υποψήφια το πράσινο κουμπί, κυρία Μόη το δεύτερο. Είναι σαφής λοιπόν η διαδικασία για σας. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ξεκολουθεί να είναι ανοιχτή η ψηφοφορία. Δεν σημειώνονται τεχνικά προβλήματα. Τώρα έληξε η ψηφοφορία. 26 ψήφοι υπέρ της κυρίας Νταντσίλα και 11 υπέρ της κυρίας Μόη. Συγχαίρω την κυρία Νταντσίλα και την παρακαλώ να προσέλθει στα έδρα του Προεδρείου. Κυρίε και κύριοι, εκλέξαμε έτσι το Προεδρείο της Επιτροπής Γεωργίας. Είναι βέβαια περιορισμένος ο χρόνος μας, διότι θα ακολουθήσει ευθύς αμέσως άλλη συνεδρίαση στην παρούσα αίθουσα. Το χρονοδιάγραμμά μας για το 2014. Στις 4 Ιουλίου λάβατε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε σχέδιο το χρονοδιάγραμμα για τις συναντήσεις του υπολείπου του έτους και αν δεν έχετε σχόλια οι παρατηρήσεις, τότε θα εγκριθεί το σχέδιο αυτό. Έχετε σχόλια? Όχι. Άρα εγκρίνεται το χρονοδιάγραμμα. Το 4 διαγράφεται. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 23 Ιουλίου εδώ στις Βρυξέλλες. Συγχαίρω και πάλι τα πρόσωπα που εξελέγησαν ως ευρωβουλευτές καθώς επίσης ευχαριστώ όλες και όλους εσάς που αποφασίσατε να γίνετε μέλη στην παρούσα Επιτροπή. Κύριε Κούσμεκ, θα ήθελα πρώτα να σας συγχαρώ κύριε Πρόεδρε για την εκλογή σας Και θα ήθελα επίσης να αναφέρω ένα σημαντικό πρόβλημα που απασχολεί τους γεωργούς και ιδίως τους πόλεμους γεωργούς τις κυρώσεις δηλαδή για το 13-14 για την υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος. Είναι αργά πλέον για οποιαδήποτε παρέμβαση, αλλά θα ήθελα εσείς και το Προεδρείο να εγκύψετε στο θέμα, διότι το πρόβλημα αυτό φύγει 36.000 γεωργούς στην Πολωνία. Οι ποσοστώσεις του γάλακτος στην Ευρώπη διέπονται από ιδιαίτερους κανόνες, οι οποίοι όμως, θα, οι προστώσεις δηλαδή, θα καταργηθούν για τα έτη 15-16. Για τα 2013-14 έτη δεν ξεπεράστηκαν οι ποσοστό στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μου φαίνεται λοιπόν ότι αυτή η επιβολή κυρώσεων σε κτηνοτρόφους δεν έχει νόημα στην παρούσα περίοδο. Θα ήθελα λοιπόν η Επιτροπή Γεωργίας να ασχοληθεί με το θέμα και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να αποφευθεί η επιβολή των κυρώσεων. Απευθύνω δε έκκληση στην Επιτροπή Γεωργίας και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθούν με το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορούμε σήμερα να συζητήσουμε θέματα ουσίας. Το πρόβλημα είναι βεβαίως σημαντικό και θα επανέλθουμε στην ε, επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας. Θα γράψουμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό. Επίσης η κυρία Χέντες Καρσία θέλει να λάβει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Απευθύνομαι στο Προεδρείο διότι πρόσφατα Είχαμε κάποιες κριτικές από το ελεγκτικό συνεδρίο για ένα ζήτημα που αφορά τα ταμεία ή τα κονδύλια για την πρόθεση του κρασιού. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσετε τον νωρίτερο δυνατόν, αν είναι δυνατόν και την επόμενη συνεδρίασή μας πριν τις διακοπές του Αυγούστου, έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο προς αντιπρόεδρος ε, ε, θα το ε, θίξει το θέμα αυτό για να δούμε τι ακριβώς ε, μπορούμε εμείς να κάνουμε μετά από αυτές τις κριτικές του ελεγκτικού συνεδρίου για να μην δέχεται επιθέσεις ο τομέας του ίνου από κάποιο άλλο θεσμικό όργανο. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ναι, θα διατυπώσουμε αυτό το αίτημα. Έχουμε να κάνουμε με αρκετά κατεπήγοντα ζητήματα. Η γραμματεία μας ε, σημείωσε το αίτημά σας. Η επόμενη κυρία Μόη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω το εξής. Ένα πράγμα μόνο. Σήμερα εσείς έχετε δολοφονήσει τη δημοκρατία. Πολύ απλά αυτό είχα να πω. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, για τη δήλωση αυτή. έλεγαν. Φλάναγκαν. Ε, άκουσα ότι δεν θα ασχοληθούμε με θέματα ουσία σήμερα, το κατανοώ αυτό. Υπάρχει όμως ένα θέμα ε, πολύ επίγον για τη χώρα μου αυτή τη στιγμή και έχει να κάνει με την εμπορία βοηδών. Υποτίθεται ότι υπάρχει μία αγορά. Όμως στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας η κατάσταση είναι τέτοια ώστε ναι, μεν μπορούμε να στέλνουμε ε, στην Ιταλία ε, τα βοηδή, δεν μπορούμε να τα στείλουμε στη Βόρεια Ιρλανδία όπως την αποκαλούν ε, κάποιοι, ε, δηλαδή κάποιες δεκάδες χιλιόμετρα πιο πέρα, ε, στον Ηνωμένο Βασίλειο. Κάτι πρέπει να γίνει για αυτό το θέμα και γρήγορα μάλιστα, διότι ναι, είναι ελαττωματική η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αν έχει κάτι καλό, ε, λίγα καλά έχει, ένα είναι ότι μπορούμε ε, να έχουμε εμπορικέ σχέσει και συναλλαγές. Ε, όχι όμως στη δική μου περιοχή. Έχουμε καρτέλ και εγκληματίες που παρεμποδίζουν την συναλλαγές και τις εμπορικές σχέσεις. Ξέρω ότι έχουμε κανόνες και νόμους, όμως εμείς δεν μπορούμε ούτε εμπορικές σχέσεις, δεν μπορούμε τα προϊόντα μας να διαθέσουμε στο εμπόριο. Κάτι πρέπει να γίνει nie możemy prowadzić dyskusji Ο πρόεδρος δεν μπορούμε να συζητήσουμε για το θέμα αυτό σήμερα δυστυχώς. Λαμβάνουμε υπόψη την δήλωσή σας. Λυπούμε που δεν έδωσε το λόγο στην κυρία Μαγκίνες. Δεν σας είδα πριν. Είστε η τελευταία που λαμβάνει το λόγο. Οι τελευταίοι έσονται πρώτοι, πρόεδρε. Και οι πρώτοι έσονται τελευταίοι να σας συγχαρώ πρώτα. αλλά έχω μια παρατήρηση. Υπάρχουν πολλά σημαντικά θέματα που έθεσαν ήδη οι συνάδελφοι. Το πρώτο θέμα που θα συζητήσουμε λοιπόν στην επόμενη συνεδρίαση είναι ένας γύρος των χωρών μελών και να δούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι στην Ιρλανδία, οι άλλοι αλλού κτλ. Να αρχίσουμε λοιπόν να συζητούμε τα πραγματικά θέματα των αγροτών στην Ευρώπη. Και καλή τύχη με την Προεδρία. Ο κύριος Ντες θέλει ακόμη το λόγο. Ευχαριστώ. Εγώ ήθελα να τονίσω ότι βεβαίως αντιλαμβάνομαι πρέπει να λήξει η συζήτηση. Κυρία Μόη, δεν σκοτώθηκε σήμερα η δημοκρατία. Σήμερα η δημοκρατία η κατήσχησε διότι η ψηφοφορία ήταν δημοκρατική. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακόμη ένας. Αυτά δεν είναι αληθινή δημοκρατία, λέει η κυρία Μόη. Κύριε Φεράντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν παρουσιάσετε το πρόγραμμά σας πριν από τις εκλογές. Εδώ δεν μιλούμε για κοινή αγορά. Μιλούμε για πάτες. Θα είμαστε παρόντες εδώ για να υπερασπιστούμε την, ε, τον γαλλικό πολιτισμό μέσα σε μια Ευρώπη αλλά όχι για να συμμετάσχουμε στα παζάρια μεταξύ απαταιώνων. Ευχαριστώ. Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε άφθονο χρόνο να συζητήσουμε και αυτό το θέμα που σας απασχολεί. Θα ασχοληθούμε με τα θέματα ουσίας την επόμενη φορά που θα είμαστε εδώ. Σας έδωσα την ευκαιρία να επισημάνετε ορισμένα επίγοντα θέματα που είναι πραγματικά και σημαντικά, αλλά θα τα συζητήσουμε και αυτά και άλλα στο μέλλον. η γραμματεία σημείωσε τα θέματα που θέσατε. Σας ευχαριστώ που με εκλέξατε και ευχαριστώ που και θα τα πούμε στις 23 Εβδόμου.